Σας ευχαριστώ. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, μου εξηγήσατε πόσο σημαντικό είναι για σας το να υπάρχει ένα αηφόρο σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη. Και μου μιλήσατε για την στράτευσή σας για ένα ευρωπαϊκό ποδηλατόδρομο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι έχουμε εργαστεί και οι δύο, έχουμε ζήσει και οι δύο από τις δύο πλευρές του σιδηρού παραπετάσματος, εγώ στην Πρατισλάβα μια εποχή όπου δεν μπορούσε ε, κανένας νέος να φανταστεί το μέλλον του μέσα στην Ευρώπη. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, έχουμε ζήσει μια ιστορική μετάλλαξη τα τελευταία 25 χρόνια και ιδιαίτερα από τον ψυχρό πόλεμο και την, ε, το διχασμό της Ευρώπης είχε πληγεί ο τομέας των μεταφορών. Και γι' αυτό προτεραιότητά μου θα είναι να ε, αντιμετωπίσω τις διαφορές, τα προβλήματα, τη ασυμβατότητες στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, όπω και εσεί, ε, ήμουν υποψήφιο και εγώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξελέγην βουλευτή. Είχα και εγώ, όπω και εσεί, την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλού πολίτε σε αυτή τη διαδικασία και έτσι γνωρίζω πολύ καλά ποιοι είναι οι τομεί τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση που του ε, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Οι πολίτε λοιπόν σε αυτέ τι συνομιλίε επιβεβαίωσαν ότι οι μεταφορές, ένα καλό δίκτυο υποδομών των μεταφορών, ένα καλώς λειτουργούν σύστημα των μεταφορών, ε, είναι απαραίτητο και έχει την ευθύνη για την ε, ανάπτυξη των διευρωπαϊκών διαδρόμων των μεταφορών η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω ότι μπορούμε με τον τρόπο αυτό να αποδείξουμε ότι πρόκειται για μια από τις καλύτερες αποδείξεις για το πόσο κοντά βρίσκεται η Ευρώπη στις μεταφορές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι μεταφορές και η κινητικότητα είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πιστεύω ότι η Ευρώπη στον 21ο αιώνα αξίζει ένα σύστημα του επίπεδου, παγκοσμίου επίπεδου των μεταφορών, εάν θέλουμε να παραμείνουμε ηγετικοί... Ε, σε ηγετική θέση ανά τον κόσμο θα πρέπει να έχουμε και περιβαλλοντικά και οικολογικά σωστές μεταφορές αλλά και ασφαλείς και σύγχρονες ε, μεταφορές και επιμελητεία. Έτσι λοιπόν η οικονομική, και καθώς η οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία αξιοπρεπών και ε, αηφόρων θέσεων εργασία είναι προτεραιότητα υπαριθμών ένα για την Επιτροπή της του... του Πρόεδρου Γιούνκερ. Πιστεύω ότι οι κοινέ μας προσπάθειες στον χώρο των μεταφορών ε, και το διάστημα μπορούν σημαντικά να συμβάλλουν στο στόχο αυτό. Ε, περιμένω λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνεργαστούμε ώστε να αναπτύξουμε το πακέτο των ε, επενδύσεων για 300 δισεκατομμύρια ευρώ με μια καινοτόμο προσέγγιση που θα σημάνει μόχλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών υποδομών με καλά σχέδια, με συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον ιδιωτικό τομέα μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε να βγάλουμε την Ευρώπη, έξω, να την Ευρώπη από την κρίση και να τη φέρουμε πιο κοντά σε ύψιστο του επίπεδου υποδομές για τον 21ο αιώνα όπως τις χρειάζεται και πρέπει αυτό να το κάνουμε ένα σαφέ όραμα. Πρέπει να ετοιμάσουμε την Ευρώπη όχι για αυτό που χρειάζεται σήμερα αλλά για αυτό που θα έρθει στο μέλλον, δηλαδή για αυτό που θα χρειαζόμαστε σε 10, 20 και 30 χρόνια στις μεταφορές. Άρα χρειάζεται να αναπτύξουμε φυή συστήματα μεταφορών, χρειάζεται να εργαστούμε σε πλήρως ε, διατροπικά, ολοκληρωμένα δίκτυα, στηριζόμενα στις νέες ε, τεχνολογίες, τις δορυφορικές και τις ψηφιακές. Χρειαζόμαστε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, τα οποία θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις να έχουν την επιλογή αηφόρων μεταφορών, ε, ειδών, τρόπων μεταφορών που θα μπορούν με ένα απλό πάτημα του κουμπιού σε NFS τηλέφωνο να ε, χρησιμοποιούν. 70% των ε, πολιτών λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν ε, σε αστικά κέντρα και ως εκ τούτου οι μεταφορές όλο και περισσότερο επηρεάζουν τη ζωή, τη ζωή τους είτε πρόκειται για την επιλογή του βαδίσματος, του ποδηλάτου, της οδήγησης ενός αυτοκινήτου ή της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα μεταφορών στηριζόμενο στις πιο καινοτόμες λύσεις που θα δώσει και στην Ευρώπη την ανταγωνιστικότητα της πάλι που θα εξασφαλίσει ε, θέσεις εργασίας, αυτό που ονομάζουμε cool jobs, ωραίες θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους και θα εξασφαλίσει σταθερότητα για, το ένα, ε, για τα 11 εκατομμύρια των εργαζομένων στο χώρο των μεταφορών που αυθουσιώνουν τη ζωή τους σε αυτό. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε από την ασφάλεια και την, ε, τις συνθήκες αποφυγής κινδύνων. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε το όραμα στο οποίο αναφέρομαι. Αναφέρθηκα στο δίκτυο των TNT το δίκτυο, τα ευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών δηλαδή, τα οποία θα πρέπει με ιδιαίτερη έμφαση να, να εφαρμόσουμε, με ιδιαίτερη αυστηρότητα, να χρησιμοποιήσουμε ε, όλους τους διαδρόμους και σκοπεύω να ξεκινήσω με τις νομοθετικές προτάσεις που ήδη βρίσκονται επιτάπητος, όπως το τέταρτο πακέτο για τους συντεροδρόμους, τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες, ε, μέτρα δηλαδή και ρυθμίσεις τα οποία πιστεύω μπορούμε να εξασφαλίσουμε σημαντική πρόοδο. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι έχω πλήρη επίγνωση των κοινωνικών ευαισθησιών και των ε, ανησυχιών σε σχέση με τα θέματα αυτά. Η πρότασή μου για να τα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα ζητήματα θα ήταν να εμπαθύνουμε στον ε, κοινωνικό διάλογο, να συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να δούμε πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τη βιομηχανία των μεταφορών, αλλά όχι εις βάρος των ε, εδρεωμένων κοινωνικών προτύπων και προδιαγραφών. Οι περισσότερε από τις θετικέ εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις μεταφορές Ευρωπαϊκής Ένωση δεν είχαν εξασφαλιστεί εάν δεν υπήρχε και ύψιστο επίπεδο ε, δικαιωμάτων των μεταφορών για κάθε είδο μεταφορών. Είμαι βέβαιο ότι αυτό αποτελεί και το κλειδί ε, ώστε να ε, εξασφαλίσουμε όπως καταφέραμε τελικά να σταματήσουν οι πρακτικές των εταιριών που είχαν να κάνουν με το overbooking ή τις αλλαγές προγράμματος και διαδρομών της τελευταίας στιγμής. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ε, ο ενιαίος χώρος των ευρωπαϊκών μεταφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε τρόπο μεταφορών και τους σιδηροδρόμους ασφαλώς με την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων όπως το RTMS για ε, συστημάτων σήματος που υπάρχουν ήδη σαν δυνατότητες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων ώστε να απαλλαγούμε από τις 26.000 διαφορετικούς εθνικούς κανόνες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του τομέα αυτού και, την χρήση, και να προχωρήσουμε στην χρήση κοινών επιχειρήσεων ε, όπως το Shift to Rail για να σχεδιάσουμε διατροπικούς σιδηροδρόμους για το μέλλον. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε έτσι αξιόπιστη παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών, ύψης της ποιότητας και ε, οικονομικές υπηρεσίες για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Και έτσι θα βοηθήσουμε και τους, ε, τον κατασκευαστικό κλάδο των υποδομών των σιδηροδρόμων. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι πιστεύω ακράδαντας το όραμα του αιωνενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων. Δεν μπορούμε να χάνουμε 5 δισεκατομμύρια το χρόνο επειδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό αέριο χώρο και ως εκ τούτου να πιέζουμε τα αεροπλάνα μας να παίρνουν πιο μακρινά δρομολόγια που κοστίζουν και περισσότερα αλλά και παράγουν περισσότερα, εκπέμπουν περισσότερα ε, αέρια ε, του θερμοκηπίου. Θα πρέπει να εργαστούμε και για την αποδοτικότητα των αδρομιών μας και για τη δυνατότητα να κοιτάξουμε, να στραφούμε προς την ε, γειτονία μας όπως η παραδείγμα τη Μέση Ανατολή όπου υπάρχει σημαντική, σημαντικός ανταγωνισμός. Πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για να μην χάσουμε την, το δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πολύ μεγάλη δουλειά μπορεί να γίνει από το Σέθαρ και τις εφαρμογές του που πιστεύω μαζί με το δυναμικό που έχουμε σε δορυφορική συστήματα μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας ε, και του εξεχρονισμού αυτού του κλάδου. Όπως γνωρίζετε η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός, ε, το μεγαλύτερο εμπορικό σύνολο στον κόσμο. Όλες δεν γνωρίζουμε, δεν θυμόμαστε μερικές φορές το 75% των μεταφορών μας ε, είτε πρόκειται για εξαγωγές είτε πρόκειται για εισαγωγές περνάνε από τα πλοία. 40% των παγκοσμίων των πλοίων όλου του κόσμου ανήκουν σε ευρωπαϊκά χέρια, σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι η μεγαλύτερη ε, διάβλη ε, θαλασσίων μεταφορών στον πλανήτη. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο και στον τομέα αυτόν. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο τομέα αυτό, όπω και άλλοι, θα εξασφαλίσει πλήρη ολοκλήρωση και διατροπικότητα μέσα σε ένα νέο ευρωπαϊκό χώρο των μεταφορών. Αυτό σημαίνει εξυγχρονισμό των υποδομών των ε, λιμένων και ένα σύστημα μεταφορών χωρί φραγμού. Πρέπει να βρούμε επίση αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη ατμοσφαιρική ρήπανση, γιατί όπου μιλάμε για ένα παγκόσμιο κλάδο οικονομία, οπωσδήποτε θα πρέπει να προχωρήσουμε και στο πλαίσιο τη Παγκόσμια Ναυτιλιακή Οργάνωση και αντίστοιχα για τι αεροπορικέ μεταφορέ τη ΙΚΑΟ, ε, των οποίων είναι και μέλη τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία λοιπόν μα από τα κέντρα αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση επίση στου εσωτερικού πλωτού δρόμου, που πολύ συχνά μπορούν να αποτελέσουν την καλύτερη λύση σχέση με τα προβλήματα τη ρήπανση, ε, του δυναμικού και τη προσβασιμότητα. Αλλά αυτό ο κλάδο ε, είναι κατακαιρματισμένο, με στόλο απαρχαιωμένο και πολλέ φορέ ε, πλωτέ οδού που δεν αξιοποιούνται όπω ο Δούναβης που είναι μόνο στο 15% του δυναμικού του. Με το πρόγραμμα Ναϊάδε τώρα μπορούμε να δώσουμε νέα πνοή σε αυτόν τον κλάδο και να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει να λειτουργήσουν καλύτερα και να εργαστούν πιο ανταγωνιστικά στο χώρο αυτό. Αν μου επιτρέπετε κυρίε και κύριοι θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το tour de monde, όπω το λέμε, αυτή την επισκόπηση με τις οδικές μεταφορές. 72% των ε, μεταφορών γίνονται με αυτοκίνητο, 45% των φορτίων ε, μεταφέρονται με φορτηγά, τεράστιος κλάδος λοιπόν και με σημαντικές προκλήσεις. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως καλύτερη οργάνωση των οδικών μεταφορών ώστε να μην συνεχίσουμε το φαινόμενο να ταξιδεύουν ένα στα τέσσερα φορτηγά μας άδεια στους δρόμους μας ενώ ταυτόχρονα χάνουμε 1% του ΑΕΠ μας ε, λόγω της συμφόρησης. Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα και ως προς την αρχή του ο Ριπένον πληρώνει για να διατηρήσουμε την, ε, τις υποδομές μας σε καλό επίπεδο και να οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά τις εργασίες μας. Πρέπει επίσης να κοιτάξουμε ε, να αναζητήσουμε έναν πιο εμβαθισμένο και συνολικό τρόπο για τις διαφορετικές εφαρμογές του συμφωνημένους ε, τρόπους όπως είναι κανόνες όπως είναι η αρχή του καμποτάς. Η πίεση προς τον κλάδο για τον περιορισμό των συμφορήσεων, της, ε, ε, της συγχωρήπανσης και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ταυτόχρονα μπορεί να ενισχύσει και την ασφάλεια. Είμαι αποφασισμένος ότι θα, θα αγωνιστώ για το θέμα αυτό γιατί πιστεύω ότι κάθε πρόοδο στον τομέα αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τον αριθμό των ε, δυστυχημάτων, των τροχιών δυστυχημάτων κάθε χρόνο. Με 26.000 ε, δυστυχήματα το χρόνο έχουμε υπερβολικά υψηλά ποσοστά. Πιστεύω απαράδεκτο Όπω όπως και για μένα και για εσά. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, δυνατότητα για συμβασμό προς το θέμα της ασφάλειας σε κάθε τρόπο μεταφορών και η Ευρώπη θα καταστεί ο πιο ασφαλής χώρος μεταφορών στον κόσμο. Είμαι πεπισμένος ότι πολύ γρήγορα θα δούμε και περισσότερα ευφυή οχήματα στους δρόμους μα που θα μπορούν να επικοινωνούν, να μιλάνε το ένα με το άλλο και να χρησιμοποιούν εναλλακτικέ μορφές ενέργειας ε, με ευρωπαϊκή ε, με ευρωπαϊκές εμβέλειε Αυτό σημαίνει βεβαίω το μέλλον για τον, οδικό, για τον τομέα των οδικών μεταφορών, αλλά για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ένα κανονιστικό πλαίσιο και ευρωπαϊκές υποδομές. Για το, και για το... Χαίρομαι λοιπόν. Βλέπω ότι συνδέονται εκ νέου το διάστημα και οι μεταφορές. Το διάστημα έρχεται πιο κοντά στους χρήστες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα επόμενα έτη θα είναι κρίσιμα για τη διαστημική Ευρώπη. Μέχρι το 2020 ο στόχος μας είναι να έχουμε τις υπεύθυνε υποδομές στο διάστημα για να δώσουμε υπηρεσίες μέσω του Γαλιλαίου και του Κοπερνίκου, Για να το πετύχουμε θα θέσουμε σε κυκλοφορία πάνω των 30 δορυφόρων τα επόμενα 5 χρόνια. Έχουμε μια ισχυρή βιομηχανική βάση, ιδιαίτερα προχωρημένη τεχνολογικά. Τα διαστημικά προγράμματα της Ένωσης θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της, θα δώσουν κίνητρα για την έρευνα και την καινοτομία και θα δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης υψηλού επίπεδου. Να μην ξεχνάμε όμως ότι κυρίως το διάστημα είναι στην υπηρεσία των πολιτών όταν χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους, όταν κάνουν συναλλαγές οικονομικές, όταν παίρνουν το αεροπλάνο, όταν βλέπουν ειδήσει για τον καιρό ή ψάχνουν το πιο κοντινό ε, εστιατόριο μέσα από το αυτοκίνητό τους, χρησιμοποιούν τις διαστημικές υποδομές. Το 7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ εξαρτάται από τις διεθνείς εφαρμογές ε, κυκλοφορίας ε, και ρύθμισης ε, από πλευρά των δορυφόρων. Βέβαια όλα αυτά είναι δύσκολα να τα πετύχουμε, ε, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Το ατύχημα το οποίο συνέβη ε, στα πλαίσια του δορυφόρου για τον Καλλιλέο τον Αύγουστο δεν πρέπει να μας απογοητεύει, αντίθετα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα αυτό και να του δώσουμε μια νέα όθηση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, οι μεταφορές είναι ένας τομέας ο οποίος φύγει τους πάντες, αφορά καλύτερα τους πάντες. Είναι ο σκελετός αν θέλετε της σύγχρονης κοινωνίας. Οι επιμελητιακές λειτουργίες και οι μεταφορές γενικά στηρίζουν κάθε μορφή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Εφόσον με επιβεβαιώσετε θα συνεργαστώ μαζί σας έτσι ώστε να, να ενισχύσουμε αυτή την ηγετική θέση της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα, να δώσουμε μια νέα όθηση στην οικονομία, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, καινοτομία να προχωρήσουμε και να ε, φυσικά προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ.